Καλησπέρα σας. Ξεκινάμε με το σημείο 11, ανταλλαγή απόψεων με τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας, ε, την οποία εκπροσωπεί η κυρία Κάρν Κέρτης, ε, υποδιευθύντρια του Τμήματος Διεθνών Προτύπων του ΑΕΛΟ. Θα μας ενημερώσει για τις συζητήσεις που έλαβαν χώρα στην Επιτροπή Εφαρμογής των Προτύπων του ΑΕΛΟ κατά τη διάρκεια της 106ης Συνόδου της Διεθνούς Διάσκεψης Εργασίας τον προηγούμενο Ιούνιο. Θα μας ενημερώσει για την κατάσταση σε ορισμένες χώρες οι οποίες μας απασχολούν τακτικά στην Επιτροπή Εξωτερικού Εμπορίου. Ε, συνεργαζόμαστε και ανταλλάσσουμε απόψεις τακτικά με την Διεθνή Οργάνωση Εργασίας. Ε, Είμαστε, χαιρόμαστε που έχουμε τη δυνατότητα να εντείνουμε ακόμα περισσότερο και να μαθαίνουμε τις επαφές μας. Ε, ειδικά σε αυτή την Επιτροπή, είναι σημαντικό να συναντιόμαστε τακτικά. Ε, σε ό,τι αφορά τον, την, ε, νομίζω ότι ε, η ανταλλαγή απόψεων για, τις, ε, για τις, των εθνών κανόνων θα εμβαθύνει τις εργασίες μας. Ευχαριστώ πολύ κύριε έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να παραστώ εδώ. Η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας δίνει ιδιαίτερη σημασία στις δικές σας εργασίες και χαιρόμαστε για την συνεργασία μας όλα τα τελευταία χρόνια. Συνεχίζουμε να στηρίζουμε τις εργασία σας για θέματα της αρμοδιότητας μας. Η δήλωση του 1998 για τις ε, θεμελιώδεις αρχές ε, ε, στους χώρους στην εργασία είναι η βάση για τη συνεργασία μας. Ε, και για την, ένα μεγάλο κομμάτι της ε, δουλειάς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ILO να προωθήσουν τα θεμελιώδη δικαιώματα, εργατικά δικαιώματα. Ε, σε ό,τι αφορά την, μάλλον η Επιτροπή Εφαρμογής των Προτύπων, δίνει ιδιαίτερη σημασία σε αυτή την δήλωση όταν συντάσσει την μεσαιρία ταξής. Η το δικαίωμα συλλογικέ διαπραγματεύσει και του συνεταιρίζεστε αποτελούν σημαντικά δικαιώματα και συζητούμε πάρα πολύ συχνά ε, το πώς ε, εφαρμόζονται οι συμβάσεις ε, επιθεώρηση εργασία ανά τον κόσμο. Τελευταία, χώρε οι οποίες δεν έχουν επικυρώσει αυτές τι συμφωνίε, αναγνωρίζουν την σημασία τους και προχωρούν λαμβάνοντας βήματα να πλησιάσουν ε, στα πρότυπά μας ε, με την προοπτική ε, να επικυρώσουν τις συμφωνίες οι οποίες ακόμα δεν έχουν επικυρωθεί. Θα σας δώσω περισσότερες λεπτομέρειες γι' αυτό αργότερα. Επιπλέον, η δήλωση του 2008 για την κοινωνική δικαιοσύνη για μια δίκαιη παγκοσμιοποίηση του ILO δίνει την ε, βάση για την αξιοπρέπεια στο, στη χώρα εργασία που καλύπτεται από ε, τον κοινωνικό διάλογο, θεμελιώδη δικαιώματα ε, και την κοινωνική αλληλεγγύη. Ε, γνώμονάς μας είναι αυτή η δήλωση προκειμένου να δούμε το πώς επηρεάζουν οι, κοινων... οι διεθνείς πολιτικές τα θέματα εργασίας. Από αυτή την δήλωση του ΆΕΛΟ, με βάση αυτή τη δήλωση μάλλον, πολλά μέλη μας ζήτησαν τη βοήθειά μας ε, για να τους στηρίξουμε στη βελτίωση αυτών των προτύπων. Το τμήμα μου ε, μπόρεσε να βοηθήσει πολλά κράτη-μέλη να συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από την συμμετοχή τους στον ILO με συγκεκριμένα και εστιασμένα ε, σχέδια. Για παράδειγμα στην Μογγολία, το Πακιστάν, τις Φιλιππίνες, την Ταϊλάνδη, την Αρμενία, το Πράσινο Κροτή, το Αλσαρβαδόρ, την Γουατεμάλα και την Παραγουάη. Επιπλέον, στο πλαίσιο του, της Συμφωνίας για την Βιωσιμότητα έχουμε κάνει σημαντική πρόοδο για να αντιμετωπίσουμε προβλήματα ε, διαρθρωτικής ακαιρεότητας και ασφάλειας του χώρου Χρειάζονται ακόμα περισσότερε προσπάθειε βέβαια ε, για να γίνουν σεβαστά τα εργατικά δικαιώματα, για παράδειγμα στον Μπαγκλαντέ ε, συνεργαζόμαστε με τα αντίστοιχα όργανα του συμφώνου ε, και, έχουμε, και εξετάζουμε καταρχήν το Μπαγκλαντές. Εκεί έχουμε εργαστεί πάρα πολύ σοβαρά ε, και έχουμε σημαντικά αποτελέσματα. Πρόσθετες συνέργειες στην Γουατεμάλα και τις Φιλιππίνες με σχέδια τα οποία στηρίζονται από την Διεύθυνση ε, Αντισιακής Συνεργασίας προκειμένου να δούμε πώς ε, οι διεθνείς συμφωνίες επηρεάζουν τα διεθνή πρότυπα είναι πολύ σημαντικό ε, αυτά τα θέματα να μένουν στη μέση διάταξη και να τα εξετάζουμε συνεχώς και τακτικά. Οι συνάδελφοί μου στο τμήμα μου ε, εργαζόμαστε στο πλαίσιο αυτού του project ε, για τη Γουατεμάλα και θα συναντηθούμε, θα πάμε και μάλλον το Σεπτέμβριο και στις Φιλιππίνες τον Οκτώβριο έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε ότι θα οικοδομηθεί συνεργασία και συνέχεια και με άλλα project. Τέλος, στην Τουρκία μετά πολλά χρόνια ε, δουλειά καταλήξαμε σε ένα ε, πρόγραμμα κοινωνικού διαλόγου επίκαιρο. Η παρουσία του ILO τόπου είναι πάρα πολύ σημαντική για να βοηθηθούν τα εργατικά συνδικάτα και να εκφράσουν τις απόψεις τους και τις ανησυχίες τους, αλλά και για να χρησιμοποιηθεί ο ILO ως συνομιλητής με την κυβέρνηση. Η Διεθνής Οργάνωση πιστεύει ότι όλα αυτά δείχνουν τη σημασία, τη συνεργασία για θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Ε, ο ILO έχει πολλούς εμπειρογνώμες, πολλή τεχνογνωσία ε, και η Επιτροπή Εφαρμογής των Προτύπων ε, αποτελεί μοχλό για τον εντοπισμό των προτεραιοτήτων προς δράση. το Διεθνής Όνος έχει ως στόχο να αξιολογεί την ε, σημασία και τις επιπτώσεις του έργου ε, που γίνεται ε, στην πράξη. Από ό,τι καταλαβαίνω θα, θέλετε, θα θέλατε να ακούσετε περισσότερα πράγματα για ορισμένες από τις περιπτώσεις οι οποίες, έχουν συζητηθεί, συζητήθηκαν μάλλον στην διάσκεψη του περασμένου Ιουνίου, καθώς επίσης και για τις δραστηριότητες του ΑΕΛΟ σε αυτές τις χώρες. Θα σας πω δύο λόγια και μετά περιμένω τις ερωτήσεις σα. Καταρχήν το Μπαγκλαντές, το οποίο συζητήθηκε φέτο στην Επιτροπή Εφαρμογής Προτύπων για το θέμα της, ε, της εφαρμογής Σύμβασης για την Ελευθερία του Συνεταιρίζεστε. Το θέμα αυτό έχει συζητηθεί και στο παρελθόν πολλές φορές στην Επιτροπή Εφαρμογής των Προτύπων καθώς επίση και το θέμα της εφαρμογή της σύμβαση της επιθεωρήσεων εργασία. Γιατί αυτά τα δύο, αυτές οι δύο σύμβασεις ε, σχετίζονται πολύ μεταξύ τους. Τα θέματα τα οποία θίξαμε και εντοπίσαμε σε ό,τι αφορά την εφαρμογή αυτών των δύο συμβάσεων καταγράφονται και στο Σύμφωνο Βιωσιμότητας στις ε, δράσεις προτεραιότητες οι οποίες περιμένουμε, τις οποίες περιμένουμε από την κυβέρνηση. Ε, ο ILO και η Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο τη τη Βιωσιμότητα πιστεύουμε ότι έχουν εργαστεί με τρόπο που είναι πραγματικά κρίσιμο για να εξασφαλίσουμε πρόοδο στο Μπαγκλαντέ. Η Επιτροπή Εφαρμογή Προτύπων φέτο ε, σημείωσε, έλαβε γνώση ορισμένων ε, θεμάτων, ορισμένων κλάδων και τομέων στι οποίε έχει σημειωθεί πρόοδος. Παρόλο ότι αυτή η πρόοδο είναι ανεπαρκή και χρειάζονται πολύ περισσότερα πράγματα να γίνουν. Ένας από τους τομείς πρόοδου, τον οποίο εντοπίσαμε, ήταν η υιοθέτηση από το Υπουργείο Εργασίας ε, ε, στάνταρ διαδικασιών για την καταγραφή Χρειάζονται ε, πρωτόκολλα και διαδικασίες επίσης για την για τις ε, ε, αθέμητες εργασιακές πρακτικές. Όλα αυτά είναι σημαντικά για να εξασφαλιστεί η ελευθερία του συνεταιρίζεστε. Υπάρχουν, παραμένουν πολλά προβλήματα. Η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή έχει δημιουργήσει μια τριμερή συμβουλευτική επιτροπή που εξετάζει, επανεξετάζει την ε, εργασιακή νομοθεσία, την εργατική νομοθεσία, συγγνώμη, και πρόκειται να προτείνει λύσεις που θα εφηγραμμίσουν ε, την νομοθεσία περισσότερο με τις συμβάσεις του ILO. Δεν έχουμε στα χέρια μας τελικές προτάσεις ακόμα. Αντιλαμβανόμαστε όμως ότι ε, ο στόχος είναι να ε, μειωθεί ο, το, ο ελάχιστος αριθμός μελών που απαιτούνται για να δημιουργηθεί ένα εργατικό συνδικάτο όμως δεν γνωρίζουμε τις τελικές λεπτομέρειες. Επιπλέον, γίνεται προσπάθεια τροπής της ε, νομοθεσίας που διέπει τις ε, ζώνες εξαγωγών και μεταποίησης. Είναι ένα από τα ε, πιο περίπλοκα θέματα τα οποία αντιμετωπίζει το Μαγκλαντές. Αυτή τη στιγμή ε, συζητείται μόνο μεταξύ της αρχής που ε, ε είναι αρμοδιευτές αυτές τις ζώνες, ορισμένους, ορισμένων ε, εξαγωγέων, εισαγωγέων, εξαγωγέων βασικά ε, και κάποιων ε, κοινωνικών οργανώσεων. Προσπαθούν να δουν το κατά πόσο το καθεστώς αυτών των ζωνών συμβαδίζει με τα διεθνή πρότυπα και ε, αυτή η, και οποιαδήποτε αλλαγή θα πρέπει να γίνει σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, ε, την εργοδοσία και τα εργατικά συνδικάτα βασικά. Γιατί αυτό θα ήταν σημαντικό προκειμένου οι τελικές προτάσεις να κινούνται προς την κατεύθυνση των ετοιμάτων ε, και των ε, παρατηρήσεων που έχει κάνει η Επιτροπή Εφαρμογής των Προτύπων του ILO. Άλλα εκκρεμή θέματα στο Μπαγκλαντές έχουν σχέση με την ε, διερεύνηση των υποθέσεων των εργαζομένων που απολύθηκαν στην κρίση στην κρίση της Ινσούλια. Ε, επίσης, ε, ε, χρειάζονται βελτιώσεις ό,τι αφορά τις ε, επιθεωρήσεις εργασίας που θα πρέπει να περιλαμβάνουν και τις εξαγωγικές ζώνες. τεχνική συνεργασία, έχουμε ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα σε, σε αυτό το θέμα με τον Μπαγκλαντές. Έχουμε προσπαθήσει πάρα πολύ να βοηθήσουμε τον Μπαγκλαντές και το Υπουργείο Εργασίας να ε, ενισχύσει τις ε, ε, υπηρεσίες επιθεώρησης εργασίας έτσι ώστε να μπορούν να εφαρμόσουν τον νόμο. Αυτή η δουλειά κινείται παράλληλα με το πρόγραμμα βελτίωσης συνθήκων εργασίας του Μπαγκλαντές έτσι ώστε να βοηθήσουμε τη λειτουργία των συνδικάτων. Ωραία, περνάω στην Καμπότζη. συζητήθηκε πέρσι στην Επιτροπή εφαρμογή Προτύπων, αλλά και φέτο. για το κατά πόσον εφαρμόζεται σωστά η σύμβαση για την ελευθερία του συνεταιρίζεστε. Η κυβέρνηση πέρσι δέχτηκε ε, μια επίσκεψη αποστολή από μέρους του ΑΕΛΟ. Έγινε αυτή η αποστολή τον Μάρτιο του 2017 και η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων που θα συναντηθεί τον Νοέμβριο και το Δεκέμβριο φέτος θα αξιολογήσει τα πορίσματά της. Η, Εφαρμο... η Επιτροπή εφαρμογή ε, Προτύπων έδωσε λίγο χρόνο στην κυβέρνηση και στους κοινωνικούς εταίρους να εξετάσουν και να μελετήσουν τις συστάσεις αυτής της ε, επίσκεψης ε, και να επανεκτιμήσουν του, το εργατικό δίκαιο καθώς επίσης και τα νομοσχέδια τα που έχουν κατατεθεί για την ρύθμιση διαφορών και για άλλα θέματα. Η κυβέρνηση έχει ζητήσει τεχνική συνδρομή από τον ILO και έχει κληθεί ε, να θεσπίσει ένα νοδικό χάρτη με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα. Ελπίζουμε θα ενημερθούν οι και θα δούμε το πότε θα αντιμετωπιστούν και άλλα εκκρεμή ζητήματα. Υπάρχει επίσης σύνδεση ανάμεσα στην, συλλογικέ συλλογικές συμβάσεις και την ελευθερία του συνεταιρίζεται αφενός και το νομοσχέδιο περί ελάχιστου μισθού το οποίο εξετάζει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση και όλα αυτά τα δύο συνδέονται με την συνδρομή του ILO. Αυτά τα νομοθετικά κείμενα θα πρέπει να ευθυγραμμίζονται με τα διεθνή πρότυπα και θα ήταν χρήσιμα προκειμένου να αντιμετωπιστούν και να επιληθούν προβλήματα ε, διαφορών που έχουν προκύψει στο παρελθόν. Στον σημερινό, η Επιτροπή για την Εφαρμογή των Προτύπων επανεξέτασε και αναθεώρησε τα θέματα της, της Σύμβασης για την Ελευθερία του συνεταιρίζεστε Υπάρχει μια διαδικασία μεταρρύθμισης της εργασιακής νομοθεσίας, όμως η κυβέρνηση του Ισημερινού πρέπει να ζητήσει τεχνική υποστήριξη από τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας για να κάνει αυτή τη μεταρρύθμιση. Είναι σημαντικές οι δυσκολίες για τα συνδικάτα του δημοσίου τομέα, συμπεριλαμβανομένης της καταγραφής και εγγραφής του συνδικάτου των εργαζομένων στον τομέα της εκπαίδευσης και υπάρχουν και συνταγματικές προσταγές και επιταγές σε ό,τι αφορά τις συλλογικές συμβάσεις και τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, όλα αυτά αποτελούν προκλήσεις για τη χώρα. Η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας με τα γραφεία που έχει στην ευρύτερη περιφέρεια παραμένει διαθέσιμη στην κυβέρνηση του ή σημερινού προσπαθώντας να την επικουρήσει σε αυτή τη μεταρρυθμιστική διαδικασία για να μπορέσει η κυβέρνηση του σημερινού να αναφέρει την επίτευξη σημαντικής προόδου στην Επιτροπή των Εμπειρογνωμόνων. Στο Ελ Σαλβαδόρι έχουν εκφραστεί ανησυχίες για το κοινωνικό εργασιακό διάλογο και την εμπλοκή και δέσμευση της κυβέρνησης ε, ε, στις συναντήσεις της με τους εκπροσώπους εργοδοτών και εργαζομένων. Η πιο πρόσφατη αναθεώρηση και επανεξέτεση της κατάστασης έγινε τον Ιούνιο, τριμερής διαβούλευση σε σχέση με τη σύμβαση αυτή, με τη συνθήκη το ίδιο είχε γίνει και πέρσι περίπου και στις δύο περιπτώσεις η Επιτροπή για την Εφαρμογή των Προτύπων ζήτησε να διοργανωθεί αποστολή επιτόπου. Η κυβέρνηση δεν είχε δεχτεί αυτή την αποστολή, τη διοργάνωση, όταν συνεδρίασε η Επιτροπή για να συζητήσει ε, την ε, τριμερή διαβούλευση και τη σχετική συνθήκη τον Ιούνιο, ωστόσο ε, αμέσως μετά έγινε η αποστολή. Και ήταν πράγματι πολύ σημαντική αποστολή επιτόπου, διότι βοήθησε την κυβέρνηση, παρέστη, ήταν, ε, κάλεσε όλους να επανεμπλακούν καλή την πίστη, να ασχοληθούν για να προσδιορίσουν κριτήρια για την αντιπροσωπευτικότητα και έτσι να μπορέσει η κυβέρνηση να συγκαλέσει ε, στο Ανώτατο Εθνικό Συμβούλιο ε, την τριμερή αυτή διαβούλευση και διαπραγμάτευση. Όλα αυτά τα θέματα τα εξετάζει και η Επιτροπή των Εμπειρογνωμόνων και η Επιτροπή για την Ελευθερία του Συνέρχεστε και του συνεταιρίζεστε στην Διεθνή Οργάνωση Εργασίας. Έρχομαι τώρα στη Γουατεμάλα, όπου τα πράγματα έχουν γίνει αρκετά περίπλοκα αυτή τη στιγμή. Η σχετική επιτροπή επανεξέτασε το θέμα της εφαρμογής της Σύμβασης για την Ελευθερία του ε, του συνέρχεστε και όλα αυτά έχουν εξεταστεί επανελειμμένως και από την Επιτροπή για την Εφαρμογή των Προτύπων αλλά και από τα διοικητικά όργανα της Διεθνούς Οργάνωσης ε, Εργασίας, διότι υπάρχουν αιτήματα για την ε, σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής. Υπάρχουν διάφορα θέματα που άπτονται όλων των τομέων στη Γουατεμάλα. Μιλούμε για την ελευθερία του συνέρχεστη, για την προώθηση των συλλογικών συμβάσεων. Ε, συλλογικές συμβάσεις σχεδόν δεν υπάρχουν στη χώρα. Μιλούμε για μέτρα επιβολή του νόμου με την επιθεώρηση εργασίας, με την προστασία έναντι των διακρίσεων και τη διακρίσεις κριτική μεταχείριση και υπάρχουν και όλα τα θέματα των αυτοχθόνων και ηθαγενών. Έχει ειδικό εκπρόσωπο η Οργάνωση εργασία Επιτόπου, ο οποίο εκπρόσωπο υπήρξε εξαιρετικά αποτελεσματικό βοήθησε ιδιαίτερω στην κυβέρνηση να περάσει τι απαραίτητε νομοθετικέ μεταρρυθμίσει σε σχέση με τη δυνατότητα και την εξουσία για την επιβολή κυρώσεων, σε σχέση με τα τμήματα τη νομοθεσία που πρέπει να μεταρρυθμιστούν και να επανεξεταστούν, να ενεθωρηθούν για τι συλλογικέ εμβάσει και για τι την ελευθερία του ε, συνέρχεστε. Μιλούμε για τον ε, αντίκτυπο του εμπορίου στην απασχόληση και στα πρότυπα της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας. Έχουμε ε, project συνεργασίας με τη Γενική Διεύθυνση Εμπορίου για να βελτιώσουμε διάφορους τομείς της Σύμβασης του 87. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια θεσμική κρίση, θα το γνωρίζετε, η οποία δεν έχει καταλαγιάσει και η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας δεν ξέρει ακριβώς ε, ποια είναι η θέση της σε σχέση με τις κυβερνήσεις που ζητούν ε, να ε, σημειωθεί πρόοδος στις εργασίες εντός των Επιτροπών Εφαρμογής Προτύπων μεταξύ άλλων. Συνάδελφός μας θα πάει στη Γουατεμάλα στα μέσα Σεπτεμβρίου για να προωθήσει όλα αυτά τα θέματα που θέτει η Επιτροπή για την Εφαρμογή των Προτύπων και για να υπάρξει ένας οδικός χάρτης για την εφαρμογή του άρθρου 26 και τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής. Έρχομαι τώρα στην Ινδία. Η Επιτροπή Εφαρμογής Προτύπων αναθεώρησε το θέμα, εξέτασε το θέμα της επιθεώρησης εργασίας και όλα αυτά παραμένουν ζητήματα αρκετά λεπτά ε, δεν έχει ζητήσει επίσημος τεχνική βοήθεια η κυβέρνηση από τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας για να δοθεί συνέχεια στα αιτήματα της Επιτροπής για την εφαρμογή των προτύπων. Βεβαίως το γραφείο ε, έχει αναλάβει ισχυρή δέσμευση και θέλει να βοηθήσει την κυβέρνηση. Το ενδιαφέρον είναι ότι η κυβέρνηση της Ινδίας έχει ξεκινήσει διάλογο με τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας για τις ε, συμβάσεις, για τις φιλογικές διαπραγματεύσεις και για την ελευθερία του συνέρχεσθε, τις οποίες δεν έχει κυρώσει ακόμα ε, το κράτος της Ινδίας. Και έχει θεσπιστεί ένα γύρο συζητήσεων με συμμετοχή της Διεθνούς Οργάνωση Εργασίας για να εξεταστεί το ενδεχόμενο μεταρρύθμιση τη νομοθεσία έτσι ώστε η Ινδία να προχωρήσει προς την κύρωση αυτών των δύο συμβάσεων τις οποίες δεν έχει ακόμα επικυρώσει. Έρχομαι τώρα στο Καζακστάν και θα ήθελα να πω ότι από ό,τι καταλαβαίνω η Επιτροπή σας το έχει συζητήσει το Καζακστάν ως θέμα και νωρίτερα σήμερα το πρωί, αν δεν απατώμε. Η Επιτροπή για την εφαρμογή των προτύπων εξέτασε το ζήτημα αυτό ε, πέρυσι, ζήτησε ε, την διοργάνωση αποστολής άμεσης με επαφές επιτόπου, η οποία έγινε πέρσι το Σεπτέμβριο και το μήνυμα ήταν αρκετά αισιόδοξο για την δέσμευση και εμπλοκή και ενεργή συμμετοχή ε, του ε, ε, Υπουργείου Εργασίας. Υπήρξε συμφωνία να προχωρήσουν προς την άρση των εμποδίων για την ύπαρξη νομοθεσίας, για την ελευθερία του συνέρχεστε και για τα συνδικάτα, τις συνδικαλιστικές οργανώσεις και για τις οργανώσεις των εργοδοτών. Γνωρίζουμε ότι υπήρξαν κάποιες περιπτώσεις, υποθέσεις ε, που έφτασαν στα δικαστήρια της χώρας σε βάρος ορισμένων μελών συνδικάτων και είχαμε διαγραφή από το καταλόγο ορισμένων συνδικαλιστικών οργανώσεων και ε, κάποιες ε, φορές που το δικαστήριο εξέτασε τον τρόπο χρηματοδότησης ορισμένων οργανώσεων. Όλα αυτά τα θέματα τα εξετάζει η Επιτροπή της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την ελευθερία του συνέρχεστη. Σε ό,τι αφορά την Επιτροπή για την Εφαρμογή των Προτύπων, ζητήθηκε ε, να, η κυβέρνηση να ζητήσει τεχνική βοήθεια και να υπάρξει μια τριμερής αποστολή υψηλού επίπεδου. Δηλαδή, μία αποστολή στην οποία θα είχαμε συμμετοχή από εκπροσώπους των οργανώσεων των εργαζομένων, εκπροσώπους των οργανώσεων των εργοδοτών και εκπροσώπους της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας και της Κυβέρνησης βέβαια. Αυτό κατά πάσα πιθανότητα θα λάβει χώρα του χρόνου η κυβέρνηση δέχθηκε να λάβει τεχνική βοήθεια το Σεπτέμβριο, αλλά όλα αυτά δεν έχουν ακόμα επιβεβαιωθεί. Και υπήρξε μια συμφωνία ενίσχυσης της συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση για την προώθηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και στον χώρο εργασίας μεταξύ άλλων. Όλα αυτά είναι ένας μοχλός πίεσης για να προχωρήσει η κυβέρνηση. Ένα από τα βασικά προβλήματα σε ό,τι αφορά τις περιπτώσεις ε, για τις οποίες έχει επιληφθεί το δικαστήριο είναι ότι ορισμένα από αυτά τα θέματα δεν υπάγονται στη δικαιοδοσία του Υπουργείου Εργασίας. Άρα οι συνομιλητές μας δεν είναι σε θέση να κάνουν και πολλά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση γιατί άλλα Υπουργεία είναι αρμόδια και όχι οι συνομιλητές μας. Παρόλο που έχει ζητηθεί η διεθνή Οργάνωση Εργασίας, εμείς δηλαδή να συναντηθούμε με τα αρμόδια Υπουργεία στη χώρα αυτή. Έρχομαι τώρα στη Μαλαισία. Εκεί μιλούμε για το θέμα της καταναγκαστικής εργασίας. Η Επιτροπή για την Εφαρμογή των Προτύπων το εξετάζει, καθώς επίσης και ε, το θέμα της Σύμβασης 98 για τις συλλογικές συμβάσεις και συλλογικές διαπραγματεύσεις. Η Μαλαισία δεν έχει κυρώσει τη Σύμβαση του 87 για την ελευθερία του συνέρχεστε. και στο πλαίσιο της TPP και του σχεδίου για τη συνέπεια για τα εργασιακά ε, θέματα είχε δεσμευθεί αυτή η χώρα να μεταρρυθμιστεί για να, έτσι ώστε το δικό της δίκαιο να ε, συνάδει με τη σήμαση του 87 και του 98 για να καταπολεμηθεί και το τράφικιν η Μαλαισία λοιπόν έχει ξεκινήσει συνεργασία με τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας πολύ πρόσφατα και ελπίζουμε ότι θα συνεχιστεί η συνεργασία μας για να ακομίσουμε τις απαραίτητες αλλαγές στη χώρα αυτή. Στη Μιανμάρ τώρα που μου είπαν ότι ε, θέλετε να την ε, σχολιάσω, να σας πω ότι παρόλο που δεν συζητήθηκε στην τελευταία συνεδρίαση, έχουμε μακρά παράδοση καταναγκαστικής εργασίας παιδιών στρατιωτών στη χώρα αυτή. Υπάρχουν διάφορα θέματα για την ελευθερία του συνέρχεσθε. Υπάρχει αδίαιρετη ανάγκη να μεταρρυθμιστεί η εργασιακή νομοθεσία, η οποία μόλις πρόσφατα προέκυψε και υιοθετήθηκε έχει ένα σχέδιο η κυβέρνηση αυτή τη, αυτή στιγμή και εμείς συνεργαζόμαστε με την κυβέρνηση της Μιανμάρ για να αναθεωρώσει την, ε, την νομοθεσία της για ε, ε, την επίλυση των διαφορών και για την τα εργασιακά. Θέλουμε να προωθήσουμε μέτρα κατά των διακρίσεων, να ενισχύσουμε τις συλλογικέ διαπραγματεύσεις. Η χώρα αυτή δεν έχει κυρώσει τη σχετική σύμβαση και άρα είναι δύσκολο να ε, ε, ε, καλέσουμε την κυβέρνηση να εντείνει τις προσπάθειές της σε αυτό το τομέα. Σε κάθε περίπτωση έχει αναλάβει δέσμευση η κυβέρνηση της Μιανμάρ να προωθήσει νομοθεσία για την ελευθερία του συνέρχεστε και αυτό θέλουμε να το στηρίξουμε με κάθε τρόπο. Η Επιτροπή για την Εφαρμογή των Προτύπων εξέτασε τι στην Παραγουάη και τη Σύμβαση για την καταπολέμηση της καταναγκαστικής εργασίας. Δίδεται τεχνική βοήθεια στην Παραγουάη για τη διατύπωση του διαθεσμικού πρωτοκόλου για το συντονισμό μεταξύ βασικών φορέων και υπηρεσιών και οργανώσεων της χώρας. Αυτό ε, το βλέπουμε σε πάρα πολλές χώρες ότι υπάρχουν θέματα που ξεπερνούν τη δικαιοδοσία του εκάστοτε Υπουργείου Εργασίας και άπτονται της πεδίου αρμοδιοτήτας και δικαιοδοσίας των εισαγγελικών αρχών των δικαστηρίων Αρχών επιβολή του Νόμου κλπ. Επομένω, χρειάζεται εκπαίδευση και του δικαστικού σώματο. Ε, είναι πολλέ οι προκλήσει που έχουν να κάνουν με τους αυτόχθονες πληθυσμούς και εμεί είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε την Παραγουάη προ αυτή την κατεύθυνση. Ω προ την Τουρκία. Είναι μια χώρα που συζητήθηκε φέτος και εξετάσαμε το θέμα αυτό ως προς τη Σύμβαση για τους εκπροσώπους των εργασομένων και φυσικά μπορώ να πω ότι το τα σχόλια για την Τουρκία δεν, δεν είχαν να κάνουν με τις απολύσεις ε, και τις πάρα πολλές απολύσεις που έγιναν μετά την κήρυξη της χώρας σε ε, κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Ωστόσο, η Επιτροπή Εφαρμογής των Προτύπων εξέτασε ε, διάφορα θέματα το ενδιαφέρον είναι ότι δεν πήρε το λόγο κανείς εκπρόσωπος της κυβέρνησης και αυτό μας εξέπληξε στην Επιτροπή Εφαρμογής των Προτύπων εντός της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας. Υπάρχει το project για το κοινωνικό διάλογο. Αυτό είναι ένα πρόγραμμα, ένα σχέδιο που είναι έτοιμο να βοηθήσει τα συνδικάτα να γύρουν τις ανησυχίες τους κάθε φορά που νιώθουν ότι... Ε, βρίσκονται στο στόχαστρο ε, ε, κάθε φορά που νιώθουν ότι μπορεί να γίνουν απολύσει ακριβώς γιατί κάποιος είναι μέλος κάποιου συνεκαλιστικού σωματείου ή άλλου. Υπάρχει ηλεκτρονική καταγραφή για τη διευκόλυνση των συλλογικών διαπραγματεύσεων και αυτό χρησιμοποιείται αυτή τη στιγμή μόνο και μόνο για να ταυτοποιηθούν ποιοι είναι μέλη των σωματείων και ε, η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας θα παρακολουθεί όλα αυτά τα θέματα εξαιρετικά στενά. Δύο λεπτά μου μένουν, θα είμαι εξαιρετικά σύντομη, στην Ουκρανία. Υπάρχει ένα πρόσφατο πρόγραμμα για την ενίσχυση των επιθεωρήσεων εργασίας με βάση τις αξιολογήσεις της Υπηρεσίας Εργασίας της Κρατικής. Η Επιτροπή για την Εφαρμογή των Προτύπων ε, έμαθε ότι δεν έχει ανανεωθεί το μορατόριο για τις επιθεωρήσεις εργασίας και άρα θα λάβουν χώρα αυτές οι επιθεωρήσεις εργασίας και αυτό το μάθαμε με χαρά. Υπάρχει και το θέμα των ημερομεστίων και των παραπώνων που έχουν διατυπωθεί στο διοικητικό όργανο της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας. Είναι ε, πολύ σημαντικό να προχωρήσει το θέμα με τα λεξιπρόθεσμα ημερομίσθια που δεν έχουν καταβληθεί αλλά και με τα υπόλοιπα θέματα της επιθεώρησης εργασίας. Και τέλος, ως προς το Βιετνάμ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει το γραφείο, τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας και υπάρχει πρόοδος, θέλουμε να βελτιωθούν οι εργασιακές σχέσεις. Όλα αυτά έχουν αποτελέσει μέρος του σχεδίου συνέπειας στο πλαίσιο της TTIP, TPP μάλλον, και θέλουμε σταδιακά να προσεγγίσουμε όλα αυτά τα θέματα και τις ελευθερίες του συνέρχεστε και σε επίπεδο επιχειρήσεων και διαφόρων φορέων. Η κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο κύρωση της Σύμβασης του 98 για τις συλλογικές διαπραγματεύσεις η συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση υπό τις παρούσες συνθήκες είναι πολύ σημαντική για τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας και περιμένω να προγραμματιστεί συνάντηση σχετική στα μέσα του Σεπτεμβρίου. Αυτά εν συντομία ήταν τα, θέμα ε, θέματα που έχουν τεθεί στην Επιτροπή για την Εφαρμογή των Προτύπων μεταξύ άλλων. Με χαρά μου να απαντήσω στις ερωτήσεις σας. Η Πρόεδρος, σας ευχαριστώ. Προτείνω να προχωρήσουμε ευθύ αμέσω στην ανταλλαγή απόψε με τους συναδέλφους. Ο κύριος Ρούας παρακαλώ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Μία ερώτηση έχω. Αλλά καταρχήν θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την τόσο λεπτομερή παρουσίασή σας. Η ερώτηση μου είναι γενική φύσεως. Στην Ολομέλεια του Ιουλίου του 2016, αφού είχαν περάσει τρία χρόνια από την τραγουδία του Ρένα Πλάζα ε, συμφωνήσαμε να ξανατονίσουμε τις δεσμεύσεις, να θυμίσουμε τις δεσμεύσεις της κυβέρνησης του Μπαγκλαντές. Να... Και ζητήσαμε η κυβέρνηση να σεβαστεί την σύμβαση του ΑΕΛΟ του 87 και όλο το εργατικό δίκαιο στις ε, ζώνες ελεύθερων συναλλαγών ε, και τις εξαγωγικές ζώνες. Στην ολομέλεια, σε μια ολομέλεια φέτος ζητήσαμε από την Επίτροπο ε, και από την κυβέρνηση του Μπαγκλαντές να μην σταματήσουν τις εργασίες τους προκειμένου αυτές οι δεσμεύσεις να γίνουν πραγματικότητα να υλοποιηθούν. Ζητούσαμε από την εκπρόσωπο του Άιλο, ε, μάλλον θέλω να ρωτήσω ε, την εκπρόσωπο του ILO, αν πιστεύει ότι ο ρυθμός με τον οποίο κινείται το Μπαγκλαντές είναι πολύ αργός ακόμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Ρουάς. Ο κύριος ε, Μάρτιν έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε την Διεθνή Οργάνωση Εργασίας για την παρουσίαση που μας έκανε. Ε, πρέπει να πω ότι ε, ακούστηκε μια λεπτομερής παρουσίαση για αρκετέ χώρε, αλλά υπάρχουν και κάποιε άλλες που θα μα ενδιαφέρουν. Εμείς στην Επιτροπή μας ανησυχούμε πολύ για την κατάσταση στη Νότιο Κορέα και ελπίζαμε ότι η αλλαγή του Προέδρου θα σήμαινε κατ' ουσίαν και αλλαγή στάσης της κυβέρνησης της ε, Νότιας Κορέας. Και θέλω να ρωτήσω μήπω η διεθνή Οργάνωση εργασία έχει έρθει σε επαφή με αυτή τη χώρα για την βελτίωση των ε, σχέσεων, των εργασιακών σχέσεων. Και κάτι άλλο θέλω να ρωτήσω. Στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ε, ακούσαμε και διαπιστώσαμε ότι υπάρχει επιδείνωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όχι μόνο στις Φιλιππίνες, σε όλες αυτές τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας. Η ΑΕΛΟ έχει διαπιστώσει να υπάρχει επιδείνωση των εργασιακών προτύπων και ε, δικαιωμάτων σε αυτές τις χώρες. Ο κύριος Σόλτς έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύρια Πρόεδρε και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω. Ευχαριστώ πολύ για αυτή την λεπτομερή παρουσίαση. Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση. Ίσως ε, την κατάσταση στις χώρες που αναφέρατε ε, πράγματι ε, να μπορεί να τη συνδέσει και με άλλες εξελίξεις. Χτες είχαμε μια συνάντηση με τους πρέσβεις ε, των τρίτων χωρών και συζητήσαμε την κατάσταση του Διεθνούς Δικαίου και των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Και ρωτώ, η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας ως θεσμός, η οργάνωσή σας θεωρεί ότι είναι απαραίτητο να συμπεριλάβει και άλλα κεφάλαια δεσμευτικά, δεσμευτικά κεφάλαια, δεσμευτικούς μηχανισμούς σε αυτά που ήδη υπάρχουν ε, για να βελτιωθεί η κατάσταση. Δηλαδή, ε, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να επιταχύνουμε τις εργασίες προς αυτή την κατεύθυνση. Θα ήθελα να ακούσω τη θέση σας και σε σχέση με αυτό θέλω να ρωτήσω ποια είναι η θέση της Διεθνής Διεθνούς Οργάνωσης ε, για τις διαπραγματεύσεις ε, που συνεχίζονται στη Γενέβη σχετικά με το κατά πόσο θα μπορούσε να υπάρξει ε, μια δεσμευτική σύμβαση για εταιρική ευθύνη. Εδώ αλλάζει, αλλάζουν τα πράγματα και αν πραγματικά επιθυμούμε μία αλλαγή, πρέπει να βρούμε τα εργαλεία τα οποία σε αυτήν την παγκόσμια λυσίδα αξιών εργαλεία που θα δείχνουν ότι δεν φτάνε μόνο οι κυβερνήσεις, αλλά και οι επιχειρήσεις, οι οποίες καλούνται να συνειδητοποιήσουν ότι πλέον υπάρχει αυτή η αλυσίδα που αφορά την οργάνωση της παραγωγής. Εγώ θα ήθελα να γνωρίζω ποια είναι η θέση της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας επ' αυτού του θέματος. Σας ευχαριστώ. Συνάδελφοι, παρακαλώ να είστε σύντομοι για να μπορέσει η κυρία Κέρτης να απαντήσει και να μιλήσει και η Κομισιόν πριν τις 4 η ώρα. Η κυρία Κίρτον Ντάρλιν, παρακαλώ. Εγώ θα ήθελα να κάνω μια ευρύτερη ερώτηση που έχει σχέση με αυτά ο Helmet. Δηλαδή, Υπάρχει τώρα συζήτηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο για το πώς μπορούμε να στηρίξουμε τα κεφάλαια της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ασχολούνται, που έχουν σχέση με τη βιωσιμότητα. Και τι θα γίνει στο μέλλον. Αυτά έχουν σχέση και με τα εποπτικά εργαλεία της ε, ΑΕΛΟ είτε με την Επιτροπή των Εμπειρογνωμών, είτε με την Επιτροπή της Εφαρμογής των Προτύπων. Πάντως, εμάς μας ενδιαφέρει να μας πείτε τη δική σας την άποψη πώς δηλαδή η ΑΕΛΟ μπορεί να ε, παίξει πιο ουσιαστικό ρόλο ε, στα κεφάλαια αυτά που θέλουμε να προσθεθούν σε διμερές επίπεδο αλλά και σε πολυμερείς προσπάθειες που καταβάλλονται. Έχω την εντύπωση ότι δεν μπορούμε να εστιάζουμε μόνο στην εφαρμογή των προτύπων, αλλά θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι η Επιτροπή αυτή είναι πολιτική και είναι πολύ δύσκολο για την ΑΕΛΟ να επιτύχει τριμερείς συμφωνίες και να προσθέσει κάποιες παραγράφους. Εγώ θέλω να γνωρίζω, όταν εγκρίνεται μία συγκεκριμένη παράγραφος, ένα συγκεκριμένο άρθρο, Τελικά τι γίνεται. Ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση στην εμπορική της ε, πολιτική ε, δεν δεσμεύεται Αναφέρεται, ας πούμε, την περίπτωση της Γουατεμάλας. Εκεί υπάρχουν ειδικά άρθρα που αφορούν στη Γουατεμάλα και παρόλα αυτά βλέπουμε ότι αυξήθηκε ε, η δυνατότητα πρόσβασης Μπάλα σε εμπορικές σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση στην αμφιλεγόμενη περίοδο. Άρα δηλαδή, ρωτώ, εσείς τι λέτε, ε, είναι συμβατή η εμπορική πολιτική με αυτούς τους στόχους βιωσιμότητας που βεβαίως ε, όλοι μας προσυπογράφουμε. Εγώ πιστεύω ότι θα έπρεπε να υπάρχει αρμονία ανάμεσα στα δύο και είχα και την εντύπωση ότι και η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας παίζει καθοριστικό ρόλο. Θέλω να ακούσω την άποψή σας επ' αυτού. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ε, θα είμαι σύντομη ε, λόγω του ότι ε, δεν έχουμε αρκετό χρόνο στη διάθεσή μας. Θα ήθελα να αναφερθώ στην έκθεση ε, της ε, ομάδας Γεωργίας της Ολλανδίας για την Ινδία. Η Ινδία είναι πολύ λεπτό θέμα και στην έκθεση αναφέρεται ότι στην Ινδία εξακολουθεί να υπάρχει σύγχρονη δουλεία, ε, χαμηλή μισθή, επικίνδυνες εργασιακές σχέσεις, ε, αδήλωτες εργασιακές σχέσεις και σε πολλές περιπτώσεις υπάρχει και παιδική εργασία, κυρίως στην εκμετάλλευση του γρανίτη. Ίσως λοιπόν εδώ θα πρέπει να δούμε λιγάκι το θέμα της επιμέλειας ε, των παιδιών. Να μας πει η ΕΛΟ τι πιστεύει από αυτού και κάτι άλλο. Αυτό που μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή είναι η εμπορική ε, συμφωνία ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το Βιετνάμ. Το 2013 σε μία μελέτη της Επιτροπής κατέστησε σαφές ότι σε αυτή την εμπορική συμφωνία θα υπάρξει μία ουσιαστική μετατόπιση Αυτή η συμφωνία, βεβαίω, μην ξεχνάτε, αφορά εκατομμύρια ανθρώπων που εργάζονται στον τομέα τη ε, κλωστεφαντουργία. Σε πολλέ ασιατικέ χώρε, ε, στα εργοστάσια υποδημάτων ε, και στα ενδυμάτων Υπάρχουν τεράστια προβλήματα. Δεν υπάρχουν ασφαλείς εργασιακές σχέσεις, δεν υπάρχουν συλλογικέ συμβάσει. Μπορείτε να μας ενημερώσετε λιγάκι τι γίνεται ακριβώς. Υπάρχουν οι συμβάσεις ε, της Διεθνούς Οργάνωσης εργασία, Πώς εφαρμόζονται στο Βιετνάμ. Ε, θεωρώ πρέπει να γνωρίζετε ότι με αυτή τη νέα εμπορική συμφωνία ε, θα πληγούν πάρα πολλοί άνθρωποι στον τομέα της ένδυσης και της υπόδησης. Η κυρία Μόσκα. Και εγώ θα ήθελα να ε, αναφερθώ ή να ευχαριστήσω για τη λεπτομερή παρουσίαση που έγινε κυρίως για τον Μπαγκλαντές και ε, γι' αυτό που ελέγχθη ότι δεν υπάρχει ουσιαστικά πρόοδος δεν υπάρχει ουσιαστική πρόοδος στο Μπαγκλαντές. Και διαρωτώ με το εξής, η εκπρόσωπος της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας ίσως μπορεί να μας εκφράσει τη δική της ε, την άποψη σε σχέση με αυτά που απασχολούν και μας, δηλαδή πώς είναι δυνατόν να αλλάξουμε μία προσέγγιση των ε, θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσέγγιση ως προς τη συνεργασία και τον διάλογο. Ε, να υπάρχουν και δυνατότητες επιβολής ε, κυρώσεων και προστήμων. Πρέπει να είναι ή δυνατόν πιο αποτελεσματική σχέση που έχουμε με τις τρίτες χώρες. Γι' αυτό λοιπόν διερωτώ με, η εκπρόσωπος της Διεθνούς Οργάνωσης μπορεί ίσως να μας πει την άποψή της επ' αυτού. Και τέλος κάτι άλλο που είναι έτσι πολύ πιο γενικό και δεν αφορά άμεσα τα θέματα τα οποία έθιξε. Ε, ε, Παρ' όλα αυτά θέλω να σας πω ότι ξέρουμε η Διεθνής Οργάνωση έχει τοποθετηθεί και για τη μελλοντική εργασία. Αυτό είναι ένα θέμα πολύ ενδιαφέρον γιατί ξέρουμε ότι πολύ συχνά οι συζητήσεις που γίνονται συνδέουν την παγκοσμιοποίηση με την ε, τεχνολογική πρόοδο, με τις εργασιακές σχέσεις και αναφέρεται ότι τα δύο πρώτα καταστρέφουν ε, στοιχεία της εργασίας. Ίσως λοιπόν μπορείτε να μας δώσετε κάποια στοιχεία για το πώς ακριβώς η Επιτροπή σας σκοπεύει να, ε, εξετάσει αυτό το θέμα στο μέλλον. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την εκπρόσωπο του ILO για την παρουσία της εδώ και για την εξαιρετική δουλειά που κάνει. Σε γενικέ γραμμέ θα ήθελα να πω το εξή. Ποιο είναι ο καλύτερο ε, τρόπο να βοηθήσουμε να βελτιωθούν οι εργασιακέ συνθήκε ε, μέσω των εμπορικών συμφωνιών και δεύτερον, ε, βρισκόμαστε σε συζητήσει για την επικαιροποίηση τη συμφωνία με το Μεξικό. Κατά την άποψή σα ποια είναι η πραγματική σημερινή κατάσταση στο Μεξικό και ποιος είναι ο, ο καλύτερος τρόπος για να βελτιωθούν οι συνθήκες στο Μεξικό επί τη ευκαιρία των διαπραγματεύσεων. Ευχαριστώ, λέει πρόεδρος. Ο λόγος στην Κομισιόν, DG Ample και DG Trade. Και μετά στην κυρία Κέρτης. Ο κύριος Ντελαγού καταρχήν, μέρος της Κομισιόν. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω την ε, υποδιευθύντρια κυρία Κέρτης να πω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεργάζεται με τον ILO στις αναπτυσσόμενες χώρες και, και πολλά από αυτά τα προγράμματα στα οποία αναφέρθηκε υποστηρίζονται χρηματοδοτικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά δεν σταματάμε εκεί. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ δραστήρια και εντός του ILO, μεταξύ των οργάνων του ILO και στην Επιτροπή Εφαρμογής των Προτύπων. 12 ε, έγγραφα παρεμβάσεις ε, Επιτροπής, ε, στην Επιτροπή αυτή για παράδειγμα, που ήταν πολύ σημαντικά και επηρέασαν, διαμόρφωσαν τις τελικές θέσεις Επιτροπής. Επιπλέον, πολλά από τα συμπεράσματα τα έχει λάβει όψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε διάφορες δράσεις Στην εξωτερική δράση, για παράδειγμα, της, ε, ε, ε της πολιτικής απασχόλησης, ε, στις εμπορικές ε, συμφωνίες και διαπραγματεύσεις, στις ε, αναπτυξιακή της πολιτική κλπ. Η, η συμμετοχή μας στην εκατοστή έκτη διάσκεψη ήταν πολύ σημαντική. 31 ε, δηλώσεις εκ μέρους των κρατών μελών τόσο στην Επιτροπή της κ. Κέρτης όσο και στη συζητήση για τα θεμελιώδη δικαιώματα στην εργασία σε ένα καινούριο πρότυπο επίσης για την ε, απασχόληση και ε, αξιότιμη, αξιοπρεπή εργασία για την ειρήνη καθώς επίσης και στην εργασιακή, μετανάστευση. Ε, όλα αυτά, όλες αυτές μας οι προσπάθειες και η συμμετοχή μας πραγματικά επηρεάζουν το τελικό αποτέλεσμα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επίσης συνεισφέρει πολύ σημαντικά στην Επιτροπή Εφαρμογής ε, των Προτύπων στη γενική συζήτηση για το μέλλον των συμβάσεων της ε, ασφάλειας του χώρου Έχουμε υποστηρίξει την καλύτερη εφαρμογή αυτών των συμβάσεων. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση ρητά έχει ζητήσει οι συμβάσει υγεία και ασφάλεια του χώρου να εξεταστούν προκειμένου να συμπεριληφθούν στον κατάλογο των θεμελιωδών συμβάσεων. Δεν έχει συμφωνηθεί αυτό από τον υπόλοιπο κόσμο, αλλά τα συμπεράσματα υποδεικνύουν ότι ο ILO θα πρέπει να εργαστεί προ αυτήν την κατεύθυνση. Οι 12 παρεμβάσει που έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για συγκεκριμένε περιπτώσει, στι οποίε αναφέρθηκα και τι παρουσίασε η κυρία Κέρτη, ε, έχουν στο το μεγαλύτερο βαθμό ε, σχέση με διάφορες εξωτερικές πολιτικές, εμπορική, εξωτερικών σχέσεων, αναπτυξιακή κλπ. Επίσης θα πρέπει να σημειώσουμε ότι ορισμένα από τα θετικά αποτελέσματα της εργασίας του ILO είναι απόρρια συνεργασιών. Για παράδειγμα, ο Καναδάς στη διάσκεψη του ILO κατέθεσε την επικύρωση της τελευταίας θεμελιώδους σύμβασης περί ε, ε, συλλογικών διαπραγματεύσεων. Η Ινδία, από την άλλη μεριά, κατέθεσε στον ΑΕΛΣΥ το μέσο για την επικύρωση της σύμβασης για την ε, παιδική εργασία. Τους πήρε 15 χρόνια για να την περάσουν. Σημαντικό λοιπόν και αυτό. Σε ό,τι αφορά τις διάφορες χώρες στις οποίες αναφέρθηκαν, οι οποίε αναφέρθηκαν. Θα ήθελα να πω καταρχήν για τον Μπαγκλαντέ. Εκεί η Ευρωπαϊκή Ένωση παρενέβη και πριν την διεθνή διάσκεψη ε, εργασίας είχαμε έρθει επανειλημμένω σε επαφή με την κυβέρνηση του Μπαγκλαντέ και είχε ζητήσει ε, δράσεις με συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα. Η κυβέρνηση μας απάντησε και η επόμενη προθεσμία για την κυβέρνηση της είναι αύριο για το ποιε τέτοιου είδου δράσει θα αναλάβει. Οι συνάδελφοι του DG Trade, ε, μπορούν να μας δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες. Σε ό,τι αφορά τη Γουατεμάλα, είναι πολύ περίπλοκο. Το παρακολουθούμε εδώ και πολλά χρόνια. Και έχει σχέση και με το κεφάλαιο της ε, βιώσιμης ανάπτυξης και εμπορίου. Καμπότζη. Έχουμε ε, εντείνει την πίεση μας σε επαφή με τις αρχές, έτσι ώστε να πάρουμε στα σοβαρά τα πορίσματα και τις συστάσεις του συστήματος ε, του ILO. Μιανμάρ, Μιανμάρ δεν ήταν στην μέση διάταξη, την αναφέρατε όμως, η Μιανμάρ είναι μια χώρα στην οποία έχουμε την πρωτοβουλία ε, ε, εργασιακών δικαιωμάτων με στόχο την επικαιροποίηση και την πρόθεση των δικαιωμάτων αυτών στην Μιανμάρ. Νότιος Κορέα, ούτε αυτή συζητήθηκε στη διεθνή διάσκεψη, όμως ε, έχουμε ήδη έρθει σε επαφή με τον πρέσβη μεταξύ δηλαδή επιτρόπου και πρέσβη και ο πρέσβης είπε ότι η νέα κυβέρνηση θα αναλάβει την επικύρωση των υπολείπων συμβάσεων του ΑΕΛΟ που δεν έχουν ακόμα επικυρωθεί. Θα το παρακολουθήσουμε πολύ στενά. Βιετνάμ. Σε δύο εβδομάδες θα λάβει χώρα ένα σεμινάριο στο Βιετνάμ για το εμπόριο και την ανεργία, έτσι ώστε να εφαρμόζονται καλύτερα ε, τα εργασιακά δικαιώματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ντεφραντσέσκη έχει το λόγο, παρακαλώ. Η κυρία Ντεφραντσέσκη, εσύ το συγγνώμη. Μπορώ να μιλήσω και πιο μπάσα. Γιατί αντί για Φραντσέσκο με λένε Μαντλέν από τη Γενική Διεύθυνση Εμπορίου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τη συνάδελφο από τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας, την Κάρεν, και τους υπολείπους για τις παρεμβάσεις τους. Θα ήθελα με τη σειρά μου να επιβεβαιώσω αυτό που είπε ο συνάδελφος από τη Γενική Διεύθυνση για την Απασχόληση. Συνεργαζόμαστε στενά για όλε αυτέ τι υποθέσει και για όλου αυτού του φακέλου. Εν ώψη τη διάσκεψη τη Διεθνού Οργάνωση Εργασία τον Ιούνιο, κάναμε πολλή δουλειά και προσπαθήσαμε να βρούμε αντίστοιχα παραδείγματα στον τομέα του εμπορίου, ε, όπως επίσης και στον τομέα της απασχόλησης. Δηλαδή, να σας δώσω κάποια παράδειγμα, παραδείγματα. Στον Μπαγκλατές νομίζω ότι έχετε δει τις επιστολές που έχουμε στείλει. Είμαστε σε στενή επαφή και επικοινωνία με τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας. Είναι οι δύο βασικές χώρες που ψάχνουμε και εξετάζουμε με το μικροσκόπιο, αν θέλετε, με το ραντάρ μας και είχαμε συζητήσεις και συναντήσεις τον Ιούλιο και στις Βρυξέλλες και στη Τάκα. Επόμενη προθεσμία είναι 31 Αυγούστου. Πρέπει το Μαγκλαντές να, απο... να απαντήσει με συγκεκριμένα βήματα ε, σε σχέση με αυτά που ζητάμε και θα πρέπει να γίνουν περισσότερα βήματα και να εξεταστούν στο πλαίσιο του καθεστώτος γενικευμένων προετοιμήσεων GSP+, εάν δεν απαντήσει το Πακλαντές και θα συμβούν τα δέοντα. Ως προς την Πατεμάλα έχουμε στείλει ήδη επιστολή προετοιμάζοντας την σύσκεψη TST που θα γίνει αργότερα εντός του 2017, μια προειδοποιητική αν θέλετε επιστολή Και το ίδιο ισχύει και για το Σαλβαδόρ. Για την Κορέα, αυτά που μαθαίνουμε είναι ότι τους ενδιαφέρει ιδιαιτέρως και το μεταφέρουν αυτό το μήνυμα στη Γενική Διεύθυνση για Απασχόληση. Στις 21 Σεπτεμβρίου θα συναντηθεί με τον αρμόδιο Υπουργό η Επίτροπος Μάλστρομ, Σεσίλια Μάλστρομ και θα είναι αυτό πολύ σημαντικό για να δούμε κατά πόσο θα έχουν αλλάξει τα πράγματα στην πράξη. Το Βιετνάμ έχει ήδη αναφερθεί, άρα για πρώτη φορά ε, πριν από την κύρωση μία συμφωνίας έχουν γίνει βήματα και έχουμε ένα σχέδιο εφαρμογής για να δούμε ποια είναι τα κενά και που πρέπει να καλύψουμε και τα εμπόδια που πρέπει να υπερπηδηθούν. Και θέλω δύο τελευταία σχόλια να κάνω. Στι συμφωνίε ελευθέρου εμπορίου τα κεφάλαια TST είναι ε, δεσμευτικά. Δεν έχουμε χρησιμοποιήσει αυτή την εξουσία, αλλά δεν θα διστάσουμε να το πράξουμε αν αυτό αποδειχθεί απαραίτητα. Και τι παραπάνω μπορεί να γίνει με τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας. Έχουμε ήδη καλή συνεργασία, η οποία έχει ενταθεί και καλό στο τελευταίο 1,5 χρόνο. Έχουμε τακτές επαφές και εντοπίζουμε όλους τους τομείς που μας ενδιαφέρουν, όχι μόνο στα του εμπαωρίου, αλλά και σε άλλους τομείς όπου μπορούμε να λειτουργήσουμε ως μοχλή άσκησης Ευχαριστώ. Δίνω το λόγο στην κυρία Κέρτης για να απαντήσει. Πέντε λεπτά παρακαλώ, όχι παραπάνω. Ευχαριστώ πολύ. Θα προσπαθήσω να απαντήσω κι εγώ γρήγορα όσο μπορώ στα πολύ περίπλοκα ερωτήματα. Ας μιλήσουμε για τις ερωτήσεις που έχουν να κάνουν με τις εκάστοτε χώρες. Τέθηκε ερώτηση για τον Μπαγκλατές. Πώς μπορούμε να κάνουμε περισσότερο και πιο γρήγορα. Ε, όπως είπαν και οι συνάδελφοι από τη Γενική Διεύθυνση Εμπορίου, και απασχόλησης. Πράγματι, οι επιστολές που ζητούν από την κυβέρνηση δεσμευμένο χρονοδιάγραμμα για την ανάληψη δράσεων αποτελούν καλό κίνητρο έτσι ώστε η κυβέρνηση να αρχίσει να εργάζεται με σοβαρότητα για τα θέματα αυτά. Τώρα, μένει ακόμα να φανεί ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Όμως, αυτό είναι ένα μέρος της διαδικασίας και είναι σημαντικό. Παραμένουν βασική δυσκολία οι ζώνες επεξεργασίας μεταπίεσης για εξαγωγές και παραμένει το βασικό ερώτημα γιατί να ισχύουν διαφορετικά πρότυπα σε αυτές τις ζώνες μεταπίεσης με προορισμό τις εξαγωγές και να μην μπορεί να μπει τοπικός εγχώριος επιθεωρητής εργασίας μέσα. Όλα αυτά μπορεί να έχουν να κάνουν με την παγκόσμια λυσίδα εφοδιασμού. Στη Νότιο Κορέα έχουμε ενημερωθεί ότι η κυβέρνηση πράγματι εξετάζει το ενδεχόμενο μεταρρύθμιση της νομοθεσία για να μπορέσει να ακυρώσει τις συμβάσεις του 87 και του 98 και να ευθυγραμμιστεί με τα δέοντα αλλά και η Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου με την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ σημαντική για αυτή τη μεταστροφή τη θετική της κυβέρνησης. Στις Φιλιππίνες ε, τα ανθρώπινα δικαιώματα, η κατάστασή τους έχει επιδεινωθεί, ωστόσο τα εργασιακά δικαιώματα δεν έχουν υποστεί τόσο μεγάλο πλήγμα. Η κυβέρνηση συνεργάζεται αρκετά με τα κινήματα για τα ε, συνδικαλιστικές οργανώσεις, γιατί άλλωστε βοήθησαν ε, τον Πρόεδρο να εκλεγεί. και ε, ε, τους ενδιαφέρει πολύ να εφαρμόσουν τα πρότυπα. Επομένως, στα διεθνή εργασιακά πρότυπα η κατάσταση δεν είναι τόσο άσχημη όσο σε άλλους τομείς, αλλά βεβαίως συνεχίζουμε την συνεργασία μαζί τους. Θα ήθελα να τονίσω επανειλημμένος αυτό που τόνισε και, ο, και η εκπρόσωπος της Γενικής Διεύθυνσης Εμπορίου, ότι δηλαδή οι παρεμβάσει της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Επιτροπή Εφαρμογής των Προτύπων είναι ζωτική, ζωτικότατη σημασία και σας καλούμε να συνεχίσετε να το πράτετε γιατί αυτό επηρεάζει την ποιότητα στη συνολική της συζήτησης που πολλές φορές ασκείται κριτική ότι είναι υπερβολικά πολιτική η συζήτηση, όμως οι σημαντικές δηλώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης βοηθούν τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας να εκπληρώσει την αποστολή της. Μου μένει ελάχιστος χρόνος και γι' αυτό θα ήθελα να πω ότι ως προς το εξής ερώτημα, ε, κατά πόσο είναι αποτελεσματικές οι κυρώσεις και είναι πιο αποτελεσματικό το μοντέλο που βασίζεται στις κυρώσεις και λιγότερο αποτελεσματικό το μοντέλο που βασίζεται στο διάλογο, να σας πω ότι η, Διεθνή Οργάνωση, η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας υιοθετεί πάντοτε την προσέγγιση του διαλόγου. Η Μιανμάρ ε, ακόμα και όταν επιβάλλονται κυρώσεις π.χ. στην Μιανμάρ, η υπομονή είναι το πιο σημαντικό δεν φαίνεται το μοντέλο που βασίζεται στις κυρώσεις να είναι πιο αποτελεσματικό. Σε κάθε περίπτωση η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας παραμένει στη διάθεσή σας να σας δώσει οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεται σε εσάς, τις εποπτικές σας αρχές για να προχωρήσετε τα θέματα που σας ενδιαφέρουν και που σας αφορούν. και θέλουμε να ενισχύσουμε τη συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση για την Απασχόληση και την αντίστοιχη για το εμπόριο. Πιστεύουμε ότι με τη συνεργεία των τριών μας θα έχουμε πιο θετικά αποτελέσματα επί τόπου. Ευχαριστώ. Η Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ και εγώ. Ευχαριστώ όλους για την ε, συζήτηση αυτή. Προχωρούμε λοιπόν στο σημείο 12 της ημερήσιας διάταξης, δηλαδή στην ε, ψηφοφορία. Να κάνουμε ένα, μια δοκιμαστική ηλεκτρονική ψηφοφορία. Έχετε όλε τι ηλεκτρονικέ κάρτε σας. Άρχεται η ψηφοφορία η δοκιμαστική. Ψηφίστε παρακαλώ για να δούμε αν λειτουργεί το σύστημα. Πρόεδρε, συγγνώμη. Uh, Έχω ξεχάσει την κάρτα μου. It's not very nice. <laughs> It's not red card, it's a blue card. Κυρία Μινέρ, θα σας καταγράφουμε, αλλά παρακαλώ πολύ να σηκώνετε το χέρι σας, τότε θα ψηφίσετε διανατάσεις χειρός. Très euh, je vous, propose de démarrer le vote. Ας ξεκινήσουμε τη ψηφοφορία λοιπόν. Έκθεση για τον προϋπολογισμό 2018, συντάκτης νομοδότης ο κύριος Μπρόγκε. Θα κάνουμε τη ψηφοφορία με δύο, σε δύο βήματα. Πρώτον, τις ε, τροπολογίες και δεύτερον το ψήφισμα. Καταρχήν ξεκινάμε με τις τροπολογίες, τις δημοσιονομικές. Τροπολογία 67. 57 υπέρ. Ε, 54 υπέρ. Κατά. Tout le monde a sa liste de vote Έχετε όλο τον κατάλογο πληροφοριών, ε, ψηφοφορία, συγγνώμη. Τροπολογία 6754, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 6751 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 6750 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 67 52 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 67 53 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 67 57 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 67 56 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 67-55 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται περνάμε στο ψήφισμα τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική πρόταση 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Τροπολογία 6 υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι απορρίπτεται. Απορρίπτεται. Ε, ηλεκτρονική επιβεβαίωση. Τροπολογία υπαρθμών 6. Ε, δεν έχω κάρτα, αλλά ψηφίζω κατά. Άρα λοιπόν δύο ψήφους θα τις λαμβάνουμε υπόψη χωρίς κάρτα. Τροπολογία. Ε, ε, απορρίπτεται. Συμβαστική 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Στην τροπολογία 14, πρώτο τμήμα, όχι, έχει καταπέσει. Δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές. Νομίζω ότι απορρίπτεται και πάλι εξακριβώνουμε, επιβεβαιώνουμε ηλεκτρονικά για το δεύτερο τμήμα της 14. Λίγη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Συμβαστική 5 υπέρ. Υπέρ, κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 21 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 22 υπέρ. Το ΕΛΚ έχει σταματήσει να ψηφίζει. Υπέρ της 22. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 23 υπέρ κατά αποχές θα ήθελα να το δούμε ηλεκτρονικά λίγη σοφορία εγκρίνεται συμβαστική πρώτη παραθυμών 6 υπέρ κατά αποχές Εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία. Ηλεκτρονικά. Άρχεται. Λίγη. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια κύριε Μπέργκε. Nous passons euh, στο σημείο 13. Πρωτόκολλο τη Συμφωνία Σύνδεση μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και των κρατών μελών τη Αφενό και τη Δημοκρατία τη Χιλή Αφετέρου για να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση τη Δημοκρατία τη Κροατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, μία και μόνο ψηφοφορία για το σύνολο. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Λίγη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια στην κυρία Ροντρίγκε Σπινιέρο. Σας προτείνω τώρα να περάσουμε στο σημείο 14 της ημερήσιας διάταξης. Όσοι πρέπει να αποχωρήσουν από την αίθουσα, παρακαλώ να το πράξουν γρήγορα. Παρακαλώ, συνάδελφοι, ε, μην καθυστερείτε εσείς που πρέπει να αποχωρήσετε. Προτείνω λοιπόν να περάσουμε στο σημείο 14 της ημερήσιας διάταξης, δραστηριότητες των ομάδων παρακολούθησης πριν από το, τις θερινές διακοπές, δύο ομάδες παρακολούθησης της Επιτροπής για το Διεθνές Εμπόριο συν συνεδρίασαν και θα θέλαμε να αξιοποιήσουμε αυτή την πρώτη συνεδρίαση μετά τις καλοκαιρινές διακοπές για να έχουμε έναν απολογισμό. Γιατί τη Μερκοσούρ, στις 11 Ιουλίου 2017 η ομάδα παρακολούθησης ΙΝΤΑ για τις χώρες της Μερκοσούρ συνεδρίασε για ανταλλαγή απόψεων για την κατάσταση των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ε, χωρών του Μερκοσούρ. Η συνάντηση έγινε με την ε, ε, βασική διαπραγματευτή, την επικεφαλής διαπραγματευτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Σάντρα Γκαγίνη. Το... Ε, και ε, η αρμόδια μας μίλησε για τον τελευταίο κύκλο των ε, διαπραγματεύσεων και τις εξελίξεις από το 2010 μέχρι και σήμερα και πιο συγκεκριμένα το τελευταίο διάστημα. Ο αρμόδιος είναι ο κύριος Σαλαφράγκα, ο αρμόδιος βουλευτής, ο οποίος μόλις τώρα μπήκε στην αίθουσα και θα περιμένω λίγο για να μπορέσω να του δώσω το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ διότι μου δίνετε την ευκαιρία να σας ενημερώσω. Θα ήθελα να ενημερώσω τα μέλη της Επιτροπής για το αποτέλεσμα της τελευταίας ομάδας monitoring παρακολούθηση των διαπραγματεύσεων ΕΕ και Μερκοσούρ. Δυστυχώ δεν βρίσκω το φάκελό μου και τις σημειώσεις μου. Όμως κάτι ξέρω για αυτό το ζήτημα και γι' αυτό θα μιλήσω από στήθους. Ε, μετά το τελευταίο γύρο διαπραγματεύσεων που έγιναν τον Ιούλιο, ε, έχει, έχει σημειωθεί πρόοδο. η βασική διαπραγματεύτρια μα μίλησε για αυτή την πρόοδο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τα μέλη των διαφόρων πολιτικών ομάδων για τη συνεργασία του και το ε, πνεύμα ε, συνεργασία που επέδειξαν και τη μόνιμη και διαρκή του παρουσία. Θα ήθελα να προσθέσω ότι οι διαπραγματεύσει προχωρούν ικανοποιητικά, είναι θετικό το πρόσημο. Την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε συνεδρίαση σχετική για το θέμα αυτό και ο επόμενο γύρο διαπραγματεύσεων θα γίνει κάποια στιγμή το Σεπτέμβριο. Πρόθεση μου είναι είναι να καλέσω τα μέλη της ομάδας μας, να καλέσω όλα τα μέλη της Επιτροπής που το επιθυμούν, να συνεδριάζουμε μία φορά το μήνα για να ανταλλάσσουμε απόψεις με την επικεφαλής διαπραγματεύτη από πλευράς Γενικής Διεύθυνσης Εμπορίου και να γνωρίζουμε επακριβώς την πρόοδο που σημειώνεται λεπτομερώς ε, σε κάθε έναν από τους τομείς ε, της οικονομικής δραστηριότητας που μας ενδιαφέρει. Δεν θα κρύψω από τα μέλη της Επιτροπής μας ότι ο στόχος έτσι όπως τον ανακοίνωσε η Επίτροπος και ο στόχος έτσι όπως τον υπέγραψαν οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων στα πρόσφατα Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, Συμβούλια είναι να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε αυτή τη διαδικασία την ακαθόδη, την επίπονη διαπραγμάτευση μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου. Αυτό το έχει πει η ίδια η αρμόδια επίτροπος ε, κυρία Σεσίλια Μάιλστρομ και ελπίζουμε ότι όλοι ε, θα μπορέσουν να δουλέψουν ε, με τρόπο ισορροπημένο, με τρόπο αρμονικό. Υπάρχουν ακαθόδη ζητήματα, υπάρχουν θέματα που δεν έχουν ξεπεραστεί. Έχουμε τη διαπραγμάτευση για την ανταλλαγή των ειδών και ε, αυτό δεν έχει ακόμα συζητηθεί και μένει να συζητηθεί και να αποτελέσει το βασικό αντικείμενο της διαπραγμάτευσης τους επόμενους τρεις μήνες του φθινοπόρου. Θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να μας στηρεί ενήμερους ανα πάσα στιγμή και θέλει να συνεργάζεται μαζί μας. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τους σκιώδεις εισηγητές και όλους όσοι ε, συμμετέχουν ενεργά στις, εργασίες, στις εργασίες και θα ήθελα να σας πω ότι την επόμενη εβδομάδα, την επόμενη πέμπτη μάλιστα, μία αντιπροσωπή αντιπροσωπεία ε, μελών της ε, Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης της Αργεντινής από όλα τα κόμματα και όλες τις πολιτικές ομάδες έρχονται και θα προσπαθήσουμε να τους συναντήσουμε από τις 9 μέχρι τις 10 το πρωί την επόμενη Πέμπτη. Υπάρχουν κάποιες τεχνικές δυσκολίες ως προς την ημερομηνία, αλλά οι προσδοκίες μας είναι μεγάλες, πρέπει να δράξουμε αυτή την ευκαιρία και θέλουμε να έχουμε ε, μηνιαία συνεδρίαση της ομάδας παρακολούθησης για να ε, παρακολουθούμε του σύνεγγυς ε, την πρόοδο της διαπραγματεύσης. Υπό αυτή την έννοια, ο Γενικός Διευθυντής Αρμόδια για θέματα εμπορίου θα πάρει το λόγο στον Ούπο για να μας ενημερώσει περαιτέρω και θα ήθελα να προσθέσω ότι έχω υπάρξει πρόοδο στα διάφορα κεφάλαια της διαπραγμάτευσης και το πιο σημαντικό για την ανταλλαγή των ειδών και την απελευθέρωση ε, την... Ε, είναι επιτάπητος έχουν γίνει συναντήσεις με αρμοδίους από την Βραζιλία, από τις αρμόδιες επιτροπές, από την Επιτροπή και το Κοινοβούλιο και φάνηκαν οι προσδοκίες όλων από αυτή τη συμφωνία. Θέλω να υπενθυμίσω τα δεδομένα και τα στοιχεία που μας έδωσε η Επίτροπος Μάλστρομ. Η συμφωνία με την Ιαπωνία θα ε, φέρει εξοικονόμηση ένα δις για τις επιχειρήσεις μας η συμφωνία με τη Μερκοσούρ θα έχουμε ε, εξοικονόμηση ε, τεσσάρων δίσως ε, από πλευράς κατάργησης δασμών. Όλα αυτά θα είναι προς όφελος των δικών μας επιχειρήσεων. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο σημαντική είναι αυτή η συμφωνία και ελπίζουμε όλοι να εργαστούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστώ πολύ. Η Πρόεδρος και εγώ σας ευχαριστώ. Αν δεν θέλει κάποιος το λόγο για το θέμα, σας προτείνω να περάσουμε τώρα στην ομάδα ε, παρακολούθησης Monitoring Group για το Ισραήλ η οποία συνεδρίασε για να μιλήσει για ε, την κατάσταση που έχει το θέμα με τη σήμαση και την ετικετοθεσία και την κατάσταση σε σχέση με τη συμμόρφωση και την αποδοχή των βιομηχανικών προϊόντων και τα σχετικά παρατήματα αυτού του πρωτοκόλου για τα, που έχουν να κάνουν με τα φαρμακευτικά προϊόντα. Πέραν από τους εκπροσώπους της Γενικής Διεύθυνσης για το Εμπόριο και άλλοι αρμόδιοι όπως της ε, Γενικής Διεύθυνσης για την Υγεία ήταν παρόντες για να συζητήσουν με τα μέλη. Θα ήθελα να καλέσω τώρα την κυρία Μαρία Αρένα να πάρει το λόγο και να μας ενημερώσει. Ευχαριστώ. Πραγματι η DigiTrade και η Διεύθυνση Υγείας ε, παρουσίασαν τα δύο θέματα. Το ένα που έχει σχέση με την ταυτοποίηση και τις κατευθυντήρες γραμμές τις οποίες έχει εφαρμόσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αφετέρου ε, την, ε, ε την εφαρμή της συμφωνίας που δεν έχει γίνει. Δυστυχώς δεν λάβαμε σημα... ε, πολύ συγκεκριμένες πληροφορίες από την Διεύθυνση Υγείας γιατί το θέμα το οποίο είχε τεθεί δεν ήταν τόσο τα φαρμακευτικά προϊόντα στα οποία έδωσε έμφαση αλλά ε, η συμφωνία ΑΚΑ, ΑΚ ε, και η εφαρμογή της ε, στα κατεχόμενα συγγνώμη, στις, ε, στους οικισμούς ε, του Ισραήλ στα κατεχόμενα. Δεν μπορούσαμε να, δεν μπορούσαμε να πάρουμε πληροφορίες ε, διότι η Επιτροπή δεν γνώριζε το κατά πόσον έχουν δημιουργηθεί εργαστήρια παρασκευής σε τέτοιου φαρμακευτικών προϊόντων εκεί στους οικισμούς. δεν έχει γίνει πλήρης αξιολόγηση των κατευθυντήριων γραμμών, τι ακριβώς επιπτώσεις έχουν στα κράτη-μέλη και το πώς, τα εφαρμόζουν, πώς τις εφαρμόζουν τα κράτη-μέλη. Εμείς ε, δώσαμε στοιχεία στην Κομισιόν για προϊόντα τα οποία είναι προφανές πως τις εφαρμοζουν τα κρατη μελη εμεις δωσαμε στοιχεια παραχθεί στους οικισμούς και που ε, διανέμονται ε, σαν να προέρχονται από το Ισραήλ και όχι από τους Ισραηλινούς οικισμούς στα κατεχόμενα. Ε, αυτά τα φαρμακευτικά προϊόντα λοιπόν μπορούν να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση με λάθος ετικέτες, με λαθασμένες και ψευδείς ετικέτες. Ευχαριστώ. Euh, Δεν θέλει κανείς να προσθέσει τίποτα γι' αυτό. Ωραία. Κάνουμε μια μικρή διακοπή πέντε λεπτών πριν περάσουμε στο επόμενο θέμα, το οποίο θα συζητηθεί και κλεισμένων των θυρών. Ε, μόλο οι βουλευτές, η βοηθή, η γραμματεία, η νομική υπηρεσία και οι υπάλληλοι των πολιτικών ομάδων μπορούν να παραμείνουν στην αίθουσα. Όλοι οι υπόλοιποι παρακαλώ πολύ να την εγκαταλείψουν. Ξαναρχίζουμε σε πέντε λεπτά.